Συγγνώμη για αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Αλλά υπήρξαν κάποια μικρά προβληματάκια με την ημερήσια διάταξη. Καθίστε παρακαλώ. Λοιπόν, ότι την έναρξη της συνεδρίασης. Λοιπόν, ένα πρόβλημα υπάρχει με το σημείο 9 στην ε, ημερήσια διάταξη. Θα ζητήσω από τον εισηγητή να πάρει το λόγο και να μας παρουσιάσει το θέμα, το πρόβλημα δηλαδή και την πρότασή του προκειμένου να την ψηφίσουμε. Πείτε, ρίξτε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Λούκα. Ίσως ε, μερικοί ε, να το συνειδητοποιήσουν ότι σήμερα το πρωί υπήρχε μια αναταραχή λόγω κάποιων ε, θεμάτων τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί στο κείμενο. Γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα που δεν καταγράφονται όπω τα έχουμε συζητήσει. Και γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ την Ολομέλεια να δεχτεί καταρχήν αυτή την έκθεση να την αποσύρουμε και να την αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση για να έχω τη δυνατότητα να μιλήσουμε με, τις ε, δύο, με τα δύο τμήματα για να το ξεκαθαρίσουμε. Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση αυτή που συνοψίζω να αφαιρέσουμε την έκθεση από την μυρίσια διάταξη και να την αναβάλουμε για την επόμενη φορά. Όπως είπα σήμερα το πρωί, είναι κρίμα που δεν προλάβαμε χτες να το συζητήσουμε. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος κατά. Εσείς θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της ομάδας μου να πω ότι θέλουμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση του εισηγητή κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ λογική πρόταση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ερώτησή μου επαναλαμβάνεται. Είναι κανείς κατά της πρότασης του εισηγητή που μας έκανε μόλις σήμερα το πρωί. Ωραία τότε πρόκειται για το σημείο int 818 που αναβάλλεται. Τώρα η κυρία Αναμποντέα παρακαλώ. Να έρθει στο βήμα εδώ, ε, στο βήμα εδώ και να μας παρουσιάσει το ΣΟΚ 625. Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση πριν υποδεχτούμε εδώ τον κύριο Σεύκοβιτς. domnule președinte avizul pe care îl voi prezenta Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω το θέμα αυτό που έχει να κάνει με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στις χώρες μέλη. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία έχει να κάνει με μια απόφαση να διατηρηθούν οι προτιμησιακοί προσανατολισμοί του 2018 για την αγορά εργασίας. Πρόκειται για προσανατολισμούς ε, σχετικά με τους οποίους είχαμε ήδη παρουσιάσει η έκθεση και η σημερινή έκθεση δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να επαναλαμβάνει τις συστάσεις αυτές. Και προσθέτουμε βέβαια και κάποια νέα στοιχεία προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας την πιο πρόσφατη εξέλιξη των νομοθετικών προδιαγραφών που έχουν στο μεταξύ εγκριθεί. Η Ευρωπαϊκή Ανακοίνωση, για παράδειγμα, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η οποία απαριθμεί κάποιες εξελίξεις όσον αφορά την αγορά εργασίας των χωρών μελών στις εκθέσεις αναχώρα που ε, καταρτίζονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης, πρόκειται και για άλλες προδιαγραφές οι οποίες έχουν να κάνουν με τον κοινωνικό πυλώνα, με την ψηφιοποίηση και με άλλες πτυχές οι οποίες δεν αναφέρονται στους προτιμησιακούς προσανατολισμούς αλλά που θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να προσθέσουμε εδώ. Στην ε, έκθεσή μας μιλάμε λοιπόν για τους προτιμησιακούς αυτούς προσανατολισμούς και ζητάμε πολύ συγκεκριμένα να τεθούν σε εφαρμογή και ελπίζουμε του χρόνου με τους κοινωνικούς εταίρους να μπορέσουμε να εκπονήσουμε και άλλους προσανατολισμούς για την αγορά εργασίας έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται όλες οι εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στο μεταξύ και προκειμένου να μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα τα οποία αναφέρονται στις αναχώρα εκθέσεις. Υπάρχουν τέσσερις ειδικέ περιπτώσεις, τέσσερις συστάσεις δηλαδή που αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Έχουμε προσθέσει στις τέσσερις συστάσεις που είχαμε ήδη κάποια νέα στοιχεία, τα οποία έχει συζητήσει η ΟΚΕ στις διάφορες ομάδες εργασίας και προσθέτουμε και ένα νέο σημείο που έχει να κάνει με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, τον κοινωνικό πυλώνα δηλαδή. Λέμε ότι διατηρούμε τις προηγούμενες συστάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία π.χ. και επαναλαμβάνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό τα κονδύλια αυτά να προσανατολίζονται περισσότερο στην ανάπτυξη ε, στην αγορά εργασίας, στις, ε, στα προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων, στην ε, ζήτηση και προσφορά, προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ των δύο. Και επίσης προτείνουμε και μεγαλύτερη ψηφιοποίηση, που θα απαιτήσει πολλές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Στους μελλοντικούς προσανατολισμούς, λοιπόν, πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η διαδικασία ψηφιοποίησης. Γενικά μιλώντας, πάντως, το μήνυμα το οποίο μεταφέρουμε με το κείμενο αυτό είναι το εξής πρέπει να ε, στηρίξουμε τους ε, εργοδότες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να περάσουμε από το Small Business Act και να πάμε ακόμα πιο μακριά. Γιατί όπως έχουν δείξει όλες οι μελέτες, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας, που δημιουργούν περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη. Αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Το Small Business Act εγκρίθηκε πριν από 10 χρόνια και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας ζητούν να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Όσον αφορά τώρα τις ικανότητες και τις δεξιότητες, προσφέρονται σε όλα τα διαφερόμενα μέρη. Πρέπει να υπάρχει σοβαρή συνεργασία, κοινωνικός διάλογος. Να λάβουμε υπόψη μας ότι οι αναχώρα εκθέσεις λένε ότι σε ορισμένες χώρες μέλη η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι κάτι απλά τυπικό και έχει ουσιαστικό. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση της νομοθεσίας και στην εφαρμογή της στις εκθέσεις αναχώρα αναφέρεται πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι κοινωνικοί εταίροι για να παγιωθεί η θεσμική πτυχή. Έπειτα, ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι κάτι που πρέπει να πρικοδοτηθεί κατάλληλα ώστε να μπορέσουν τα δικαιώματα αυτά στην ουσία να τηρούνται και όχι μόνο στα λόγια. Υπάρχουν τώρα και κάποιες τροπολογίες. Θα αναφερθούμε σε αυτές στη συζήτηση. Πάντως ευχαριστώ τη Γραμματεία για τη στήριξή της όταν εκπονήσαμε την έκθεση αυτή, αλλά και στα μέλη της ομάδας εργασίας που βοήθησαν πολύ. Μία συνεδρίαση είχαμε και δεν είχαμε πολύ χρόνο για να εκπονήσουμε την έκθεση αυτή, αλλά χάρη στην εργασία όλων τα καταφέραμε να προλάβουμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Thank you so much,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 Iš tikrųjų, noriu Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην συντάκτρια αυτής της γνωμοδότησης και σε ολόκληρη την ομάδα που επεξεργάστηκε την έκθεση. Εγώ δεν ήμουν μέλος αυτής της ομάδας, αλλά Εκτιμώ την ε, γνωμοδότηση αυτή την οποία και διάβασα. Ιδιαίτερα εστίασα στην πρόταση να συμπεριληφθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η Κοινωνική Εταίρη και τη σύσταση για αύξηση των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, μιλάμε όλο ένα και περισσότερο για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο, αλλά θα ήθελα να τονίσω κάποιες πτυχές οι οποίες δεν ε, αναφέρθηκαν στην γνωμοδότηση. Μιλώντας για τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, πιστεύω πως είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί μια αναφορά στην ε, πρόσφατα εγκριθήσα οδηγία περί ισορροπίας μεταξύ εργασίας εργασιακής ζωής μάλλον και ε, προσωπικής ζωής. Είναι μια ε, οδηγία που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε ένα σχετικό δίκτυ ή κριτήριο ε, καθώς είναι σημαντικό όσο και η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ των φύλων. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το θέμα της συμβουλής και της καθοδήγησης για την ε, πρόοδο στη σταδιοδρομία του εργαζόμενου, δηλαδή τι θα χρειαστεί η αγορά εργασία στο μέλλον. Για παράδειγμα, ο τομέα της φροντίδας ε, και της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να ε, προσφέρουμε καθοδήγηση στους νέους που αναζητούν προοπτικές. Σας ευχαριστώ. Η Τατιάνα Βαμπρόσκινα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Άννα να την ευχαριστήσω για την ευελιξία της και το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο εργάστηκε. Εγώ δεν ήμουν στην ομάδα εργασία, αλλά υπέβαλα τροπολογίες και έγιναν δεκτές. Επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να, να σας ε, μάλλον επενέσω γιατί δεν μιλάτε μόνο για την ποιότητα της παιδείας αλλά και για τη σημασία που έχει για τους ε, δασκάλους και τους μαθητές να προωθούν τις αξίες όπως ανοχή, δημοκρατία, ε, ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό πρέπει να ε, ενταχθεί στην εργασία μας και μέσα στις γνωμοδοτήσεις μας. Εκ πρώτης όψεως δεν είναι άμεσα σχετιζόμενο, ωστόσο ευχαριστώ που το συμπεριέλαβες. Ευχαριστώ Τατιάνα. Ρενέ Μπιλέβενς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Λέω κύριος Μπιλέβενς. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, έκθεση με την οποία συμφωνώ, αλλά έχω μια παρατήρηση για το σημείο 2-4. για κάποια στοιχεία που πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Φυσικά και είναι σημαντικό να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση αλλά εγώ από τις ασφάλειες έχω μάθει ότι είναι εξίσου σημαντικό η δυνατότητα προσαρμογής του εργαζόμενου. Αυτό είναι κάτι όλο και πιο σημαντικό και θα είναι όλο και πιο σημαντικό με την εξέλιξη της αγοράς εργασίας που διαπιστώνουμε. Οπότε θα ήθελα να υπάρχει και αυτό. Γιατί λέει ότι πρέπει να υπάρχει καλή προετοιμασία, αλλά θα ήθελα και αυτή η πτυχή να υπογραμμιστεί εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σοφία Ρετζέκερ τώρα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την γνωμοδότηση η οποία συζητήθηκε σε βάθος ε, στο τμήμα μας και είναι πολύ καλό το ότι οι τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί έγιναν δεκτές. Ε, θέλω όμως να επισημάνω ένα θέμα το οποίο είναι ακόμα ανοιχτό, ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ψηφίσουμε και αφορά στα συμπεράσματα και μετά στην ε, περίληψη. Καταρχήν, το θέμα δεν είναι να έχουμε κατά νου μόνο τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, προφανώς και πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενισχυθούν ε, και γι' αυτό το λόγο ζητάμε πραγματικές επενδύσεις. Όμως, στο σημείο 1.4 επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να περιστούμε μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το σημείο αυτό να παραμείνει στα συμπεράσματα γιατί ε, για μένα το να προβάλλονται τόσο πολύ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, αυτό αφήνει ένα τεράστιο περιθώριο ερμηνεών και ως εκ τούτου ε, εδώ υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι να προκύψει διακριτική μεταχείριση για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και για τους απασχολούμενους. Ως εκ τούτου εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω αλλά και να ερωτήσω την εισηγήτρια κατά πόσο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την γενικότερη αυτή η συζήτηση για να διευκρινίσουμε αυτήν την αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος, αλλά όχι ίστατος, έσχατος, ο κύριος Μένε. Ευχαριστώ καταρχάς πολύ την συγγήτρια για την αναζήτηση των συμβαστικών λύσεων. Εγώ θα μιλήσω για τις επενδύσεις γιατί θα ήθελα να πω ότι η προσέγγιση που προτείνει η έκθεση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή είναι σχετικά περιοριστική. Εξηγεί την αδυναμία των επενδύσεων λόγω του μεγάλου διοικητικού φόρτου και την σχετική λειτουργία του κράτους. Νομίζω πως είναι ένα στοιχείο αλλά μεταξύ άλλων Εμεί συνήθως στην Επιτροπή μας είπαμε ότι δεν είμαστε εχθρικοί στον φόρτο το διοικητικό, αλλά στον απεριτό διοικητικό φόρτο και αυτό τα αλλάζει όλα. Ε, θα πρέπει καλύτερα λοιπόν να νομοθετούμε. Η βασική μου όμως, το βασικό μου πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν αμφισβητεί την, χρηματο... την, την ε, ε, προδιαγραφεί την μετοχική που υπάρχει και επικρατεί αυτή τη στιγμή. Και εξηγώ, η αξία που δημιουργεί μια επιχείρηση στην ουσία ε, πάει στους μετόχους. Αυτό σημαίνει πως παραμελούνται οι επενδύσεις. Σε αυτή την περίπτωση το κεφάλαιο είναι περισσότερο κόστος παρά για την επιχείρηση και σας παραπέμπω σε μια μελέτη που έγινε από την ε, μια ομάδα ενό Γαλλικού Πανεπιστημίου και θα σας στείλω την παραπομπή, την αναφορά. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν πάνε αρκετά χρήματα ούτε στην έρευνα και ανάπτυξη, ούτε στις επενδύσεις και γι' αυτό και εξηγεί και τις δυσκολίες που έχουν οι εργαζόμενοι για να προσαρμοστούν κάθε φορά στις νέες ε, τεχνολογίες. Επίσης, ξεχνάμε στη ζωή να μιλήσουμε για το ρόλο της προηγούμενης συζήτησης και αιτήματο από πλευράς των εταιρεών. Οι μισθοί προχωρούν πάρα πολύ αργά και πολύ ισχνά σε σχέση με την πρόοδο της παραγωγικότητας και αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, ε, μου μένουν δύο δευτερόλεπτα και πρέπει να το πω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει το, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα, οι ελλείψεις του για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των εταιρεών και των εργαζομένων κείμενο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια που δέχτηκε τις ε, τροπολογίες μας και που μπόρεσε να φτάσει σε ε, συμβιβαστικές λύσεις. Η Άννα για να ε, ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν να, θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά το θέμα της ισότητας των φύλων και όλα αυτά τα θέματα που θέλετε να μπουν στην έκθεση, να σας θυμίσω ότι έχουμε ένα περιορισμό όσον αφορά το μάκρος της έκθεσης. Χρειάζεται και να μειώσουμε στο μισό την αρχική ε, έκθεση για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στο πλαίσιο και γι' αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε να αναφέρουμε όλες αυτές τις πτυχές αλλά το είπαμε ρητά και το ξαναλέμε ότι συμφωνούμε με τις προηγούμενες εκθέσεις της ε, ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όταν μιλάμε για τις πολιτικές επασχόλησεις και θέλουμε αυτές να εφαρμοστούν πλήρως. Στην ε, σύνοψη αναφερθήκαμε λοιπόν σε αυτές τις προηγούμενες ε, γνωμοδοτήσεις όπου ρητά αναφέρονται όλες αυτές οι πτυχές και έχουμε και συμπεράσματα σχετικά. Και όσον αφορά την δυνατότητα προσαρμογής, ε, τα είπατε ότι ζητάμε από τους εργαζόμενους, έτσι φαίνεται, να προσαρμόζονται σε ό,τι τους ζητάμε. Ε, όχι, προσαρμόσαμε την ε, τροπολογία αυτή, αυτή την παράγραφο, προσαρμογή στους τομείς της ψηφιοποίησης που θα επιφέρουν πολλές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Χρειάστηκε λοιπόν να αλλάξουμε τη λέξη προσαρμογή ε, στο ε, στην προσαρμογή προς τις νέες τεχνολογίες. Όχι προσαρμογή σε συνθήκες επισφαλούς εργασίας. Γι' αυτό κάναμε αυτή την τροπολογία. Και όσον αφορά την πρόσβαση σε ε, χρηματοδότηση και αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει καλύτερα να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα για να έχουν πρόσβαση, να βρουν πρόσβαση μάλλον σε τραπεζικά δάνεια αλλά και στους ευρωπαϊκούς πόρους και γι' αυτό και η σχετική συμβιβαστική πρόταση ε, ε το τόνισε αυτό. και έπειτα ε, στο, για την αρχή του ότι ε, ξεκινάμε από μικρά προγράμματα και μετά προχωράμε και αυτό το έχουμε πει σε πολλές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Ε, είπαμε πως πρέπει να στηριχτούν οι μικρομεσαίες δίνοντας ένα παραπάνω βήμα σε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται για αυτές τις επιχειρήσεις να, να, να ενεργήσουμε δε πρώτα σε μικρή κλίμακα. Το 99% των εταιριών είναι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, δηλαδή θα δημιουργηθούν ε, δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγορά εργασίας ε, λόγω αυτής της αρχής του να προχωράμε με μικρά βήματα. Αυτό υπάρχει ήδη. Πάμε λοιπόν τώρα στις τροπολογίες. Έχουμε την υπαριθμόν 1 στο, για το 2-3. Εδώ έχουμε συμβαστική πρόταση και θα ήθελα παρακαλώ η Άννα να μας παρουσιάσει την ε, συμβαστική αυτή πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται ε, για μια πολύ απλή συμβαστική πρόταση. Εδώ γίνονται αποδεκτές οι προσθήκες με την ε, σημείωση ότι το insecurity διαγράφεται. Κατά τα άλλα, αυτή η τροπολογία γίνεται δεκτή, το διαγράφει το insecurity, ανασφάλεια. Και βλέπετε ε, το 3-4 εξετάζει αυτό το θέμα. Ως εκ τούτου ε, γίνεται δεκτή τροπολογία, αλλά διαγράφεται η ανασφάλεια, το insecurity. Αυτό, αυτή είναι η πρότασή μας. Ε, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο που να διαφωνεί. Λέει ο Πρόεδρος, από ό,τι βλέπω δεν διαφωνεί κανείς. Ως εκ τούτου η συμβαστική πρόταση γίνεται δεκτή και περνάμε στην τροπολογία 2 για το 2-4. Γίνεται δεκτή τροπολογία από την εισηγήτρια. Διαφωνεί παρακαλώ κανείς, από ό,τι βλέπω όχι η 3 για το 311 εκεί υπάρχει συμβαστική πρόταση και θα ήθελα να παρακαλέσω την εισηγητήρα να την παρουσιάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μας συμβαστική πρόταση χωρίζεται σε τρία τμήματα. Ε, για το πρώτο τμήμα θέλω να πω ότι η πρόταση δεν γίνεται δεκτή, αλλά διατηρούμε την αρχική διατύπωση της ε, τοποθέτησης και αυτό που προτείνουμε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δημοσίευσε ήδη μια ανακοίνηση και ε, σε αυτό το κείμενο το προστίθετο 2019 και το καθεξής αυτό το δέχτηκαν και οι συντάκτες. Δεύτερον, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ε, τροπολογία των ε, ε, συντακτών γίνεται δεκτή με δύο προσθήκες. Η πρώτη προσθήκη είναι ότι καταβάλλονται προσπάθειες ε, και έχει ήδη επιτευχθεί η πρόοδος όσον αφορά το θέμα πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτό μπορέσαμε να το διαβάσουμε και στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Και δεύτερον, η πρόσβαση είναι πιο δύσκολη για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί αυτές δεν έχουν τόσο εύκολη, πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Και δεχόμετα την ε, τροπολογία με δύο προσθήκες. Συγκεκριμένα ήδη έχουν ε, καταβληθεί προσπάθειες ε, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πρόσβαση. Και το τρίτο θέμα στην προσθήκη ε, των συντακτών, αυτό το δεχόμαστε και εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία λοιπόν. Είναι κανείς κατά όλες αυτές τις προσπάθειες συμβασμών. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Γίνεται αποδεκτή με το συμβασμό η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 3-4. Τη δέχεται η συγκήτρια. Είναι κανείς κατά. Όχι. Αποδεκτή. Τροπολογία 5. Για το 3-2-1. Τη δέχεται η συγκήτρια. Είναι κανείς κατά. Αποδεκτή. 6 2-3-6, 6 αποδεκτή από την εισηγήτρια. Είναι κανείς κατά. Όχι. 7. 3-2-7 αποδεκτή από την εισηγήτρια. Είναι κανείς κατά. Αποδεκτή. 8 στο 3-3-1. Αποδεκτή η τροπολογία. Είναι κανείς κατά. Πολύ ωραία. Δεκτή λοιπόν. Η υπαριθμόν 9, 363, η τροπολογία δεκτή. Ε, διαφωνεί κανείς παρακαλώ. Εγκρίνεται, δεκτή. Η 10. Για το 1-2 η τροπολογία είναι δεκτή, διαφωνεί κανείς. Δεκτή η 11. Για το 1-4 απορρίπτεται η τροπολογία. Παρακαλώ λοιπόν ε, να παρουσιάσετε την τροπολογία, μετά θα τοποθετηθεί η συγγήτρια και μετά θα ψηφίσουμε. Και ποιος θα παρουσιάσει παρακαλώ την τροπολογία για το 1-4, παρακαλώ εσείς. Η Σοφία. Νομίζω ότι το είπα ήδη στην παρέμβασή μου ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις και ενδέχεται αυτή η αρχή να ε, αναφέρεται και σε άλλες τοποθετήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναφέρεται και εδώ μία τοποθέτηση για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Παρόλα αυτά, για μένα το αίτημα αυτό ε, είναι λίγο αμφίσιμο γιατί μπορεί να προκύψουν ε, μειονεκτήματα για την απασχόληση. Αν δούμε λοιπόν τη διατύπωση του 1.4, η πρώτη μισή πρόταση αρκεί για να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πούμε χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ε, και διαρθρωτικά μέτρα τα οποία <clears throat> μπορούν να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δεύτερη μισή πρόταση θα διαγραφεί με αυτήν την τροπολογία και νομίζω ότι παρόλα αυτά όμως τοποθετούμεθα σαφώς ε, υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παράλληλα μειώνουμε τον κίνδυνο να υπάρξουν παρερμηνίες. Ευχαριστούμε πολύ Άννα, λέει ο Πρόεδρος, η Άννα μάλλον. Ε, Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ, δεν το δέχομαι αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να εκπέμψουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι αποδέκτες ε, να κατανοήσουν ότι είναι απαραίτητο να γίνει άλλο ένα βήμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για τον επιχειρηματικό κόσμο. Ως εκ τούτου, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτό είναι ε, ένα συμπέρασμα, αλλά είναι για το 1-3 της γνωμοδότησης εκεί που γίνεται λόγος για την αναθεώρηση ε, της ε, πράξης ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό έχει γίνει δεκτό από την ΟΚΕ και πρέπει να επενθυμίσουμε ότι έχουμε συμφωνήσει να περάσουμε στην πράξη. Εγώ λοιπόν ε, θα ήθελα να κάνω έκκληση στα μέλη της ε, Επιτροπής μας να δεχτούν τη δική μας ε, διατύπωση έτσι ώστε να έχουμε μία πάγια πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι ώστε να διατηρηθεί αυτή η πρόταση στο σημείο 1 1-4. Ευχαριστούμε Άννα. Λέω Πρόεδρος, ως εκ τούτου ψηφίζουμε για την τροπολογία που απορρίπτει η συγκήτρια. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Le vote est clos. Λοιπόν, ψηφίσαμε. 217 ψήφισαν, 117 υπέρ, 85 κατά, αποχές 15. Η τροπολογία γίνεται δεκτή. Τελευταία τροπολογία, η 12. Δεκτή η τροπολογία. Διαφωνεί κανείς, υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί, παρακαλώ. Από ό,τι βλέπω όχι δεκτή η τροπολογία. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για την απασχόληση της κυρίας Άννα Μποντέα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Le 211... Πέρες. 111, 211 υπέρ, 3 κατά, 10 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Λοιπόν, περιμένοντας τον ε, Επίτροπο, σας προτείνω να εξετάσουμε τα διάφορα. Έχετε πάρει στα γραφεία σας ένα χαρτί σήμερα το πρωί που λέει ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη συμμετοχή στα διάφορα όργανα. Στα αγγλικά συνεχίζω. Τόνι Βίνταν, Κροατία, αντικαθιστά τη Λίδια Πάλιβετς, επίσης από την Κροατία, ως μέλος του Προεδρείου από 1η Ιουλίου 2019. Θα υπάρξει τελική αλλαγή στην Επίτροπη Όντι επίση. Φεραίρα Πορτογαλία αντικαθιστά όλο Ρορέντσι Πλωσιάνο που είναι μέλος του τμήματος 1 από τη Ρουμανία στην Επιτροπή Audit. Και υπάρχει επίσης και αλλαγή όσον αφορά τη συμμετοχή του τμήματος. Η κυρία Καξέρα, την Ουγγαρία, φεύγει από το τμήμα 10 και πηγαίνει στο τμήμα ΝΑΤ. Είναι κανείς κατά? αυτών ε, των ε, αλλαγών των νέων μελών στα διάφορα σώματα. Ωραία, ομόφωνα εγκρίνονται οι αλλαγές αυτές. Και χρειάζεται να εγκρίνει η Ολομέλεια την εντολή της διαδικασίας του πάνελ και ζητούμε το σώμα να εγκρίνει την επέκταση της εντολής μέχρι 24 Σεπτεμβρίου του 2019 για να υπάρξει τροποποίηση των ε, εφαρμοστικών διατάξεων. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Ωραία. Τελειώσαμε τέσσερα λεπτά πριν φτάσει ο Επίτροπος. Μην φύγετε. Μικρή διακοπή, αλλά μην βγείτε από το ημικύκλιο γιατί δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο όταν εκείνος αφιχθεί. Υπότιτλοι Authorwave Salut.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 Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που καθόσαστε στις θέσεις σας και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω και πάλι εδώ στην Ολομέλειά μας τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς. Αγαπητέ Μάρος, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ και πάλι. Και μάλιστα όχι μόνο επειδή είσαι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, αλλά επίσης επειδή στις δύο θητείες που έχεις σκίσει ως επίτροπος αρχικά είχε στις θεσμικές υποθέσεις και τις σχέσεις μαζί μας, τώρα έχει την ενέργεια. Ήσουν λοιπόν πάντα πάρα πολύ ανοιχτός, πάντα ερχόσουν να μας δεις, να μιλήσουμε, να μας ακούσεις και να λάβεις υπόψη σου τα επιχειρήματά μας. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσω ότι από τότε που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας ως αντιπρόεδρος, έρχεσαι κάθε χρόνο και συζητάς μαζί μας αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα της Ενεργειακής Ένωσης. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα στην εντολή της ε, Ευρωπαϊκής αυτής Επιτροπής, της οποίας η θητεία ολοκληρώνεται. Είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτό, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δικιά σου αποφασιστικότητα και τις ικανότητες τις διπλωματικές, έτσι ώστε να τα καταφέρεις όλοι να συμφωνήσουν για να πετύχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ελπίζουμε επίσης να επιστρέψεις για τρίτη εντολή ως Επίτροπος και η νέα ομάδα των επιτρόπων να οριστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ξέρουμε ότι γίνονται συζητήσεις στο Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ, ίσως αύριο το πρωί, τα πράγματα να είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. Πάντως ελπίζουμε οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων πολύ σύντομα να καταλήξουν σε αυτή την σημαντική συμφωνία για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επανεκκίνηση. Ε, πότε βρεθήκαμε στην Πρατισλάβα ήτανε, τον Οκτώβριο του 2016 υπό Σλοβακική Προεδρία και εγώ ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Αρμόδιας ε, για την ενέργεια και είχαμε συζητήσει μαζί και είδαμε πόσο καλά μπορέσαμε να συνεργαστούμε για κάτι το οποίο πάντα βρισκόταν στην καρδιά της εντολής σας. Δηλαδή όχι μόνο να κάνουμε σημαντικά βήματα μπροστά προς την κατεύθυνση της Ενεργειακής Ένωσης, αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά αυτής της μετάβασης, αυτής της αλλαγής. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι τόσο σημαντικό όπως είναι η Ενεργειακή Ένωση, αν δεν έχουμε μαζί μας και τους πολίτες. Αλλιώς κινδυνεύουμε να αποτύχουμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ε, τώρα για τις διαφορές θέσεις, ανακοινώσεις, προτάσεις, δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι δικιά μας η Επιτροπή έχει προτείνει σε όλες αυτές τις ανακοινώσεις ε, κλπ. Να μην τα πω εγώ, αυτά τα οποία θα μας παρουσιάσετε εσείς τώρα, γιατί ξέρω ότι συμπίπτουν οι απόψεις μας απόλυτα. Δύο πράγματα όμως θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδο τα τελευταία πέντε χρόνια. Όμως ακόμα παραμένουν πολλά. Ίσως έχουμε καταλήξει στο πλαίσιο, αυτό όμως που χρειάζεται τώρα είναι να μπούμε στο περιεχόμενο, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλές διαφορές. Δεν χρειάζεται να έχουμε βέβαια ένα και μοναδικό δρόμο να ακολουθήσουμε όλοι, μπορεί ο καθένας να ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους, αλλά να πηγαίνουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Οπότε Πιστεύω, φοβάμαι ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά από αυτό. Το βασικό που θα συζητήσουμε σήμερα δεν είναι τόσο να αξιολογήσουμε το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Ποια είναι η στρατηγική για την μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της κλιματικής ουδετερότητας για το 2005 είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος και όλοι συμφωνούν με αυτόν. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι η νέα φιλανδική κυβέρνηση αποφάσισε νωρίτερα να πετύχει αυτό το στόχο, το 2035. Σε λίγες μέρες θα αναλάβει η Φιλανδία και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε ίσως να μπορέσει να πιέσει περισσότερο προς την κατεύθυνση του στόχου αυτού. Παραμένουν όμως πολλά ζητήματα για το μέλλον. Πρώτον, οι φιλοδοξίες αυτές που έχουν καθοριστεί φτάνουν για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των ημερών. Δεύτερον, πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ώστε οι πολίτες πραγματικά να βρεθούν στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο πώς θα πετύχουμε ώστε πολλές επιχειρήσεις, πολλές έχουν ε, ήδη δεχτεί τις αλλαγές αυτές, αλλά πώς θα καταφέρουμε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, πώς οι πολίτες θα δεχτούν αυτές τις αλλαγές και πώς θα βοηθήσουμε τοπικά είτε κάποιες περιφέρειες είτε κάποιους, κάποιες ομάδες πολιτών που φοβούνται πάρα πολύ την μετάβαση αυτή να μπορέσουν να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να καταλάβουν ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία και έτσι να συμμετάσχουν στις αλλαγές αυτές με προθυμία. Θα σας δώσω το λόγο λοιπόν, γιατί εσείς είσαστε ο κύριος ομιλητής μας σήμερα το πρωί και δεν θέλω να σας αντικαταστήσω όπως καταλαβαίνετε. Απλώς επαναλαμβάνω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο σας, τις προσπάθειές σας. Στηρίζουμε τόσα κάνετε. Και όσο περισσότερα κάνετε, τόσο περισσότερο και εμείς θα σας στηρίζουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητέ Λούκα, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι. Είναι αλήθεια ότι περνάει γρήγορο καιρός και Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλέ συνεδριάσει σα. Ε, θα ήθελα να φερθώ ιδιαίτερα στο θεματολόγιο που έχουμε επεξεργαστεί από κοινού και να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τη Επιτροπή για το γεγονό ότι ε, τις συζητήσεις που γίνονται εδώ στις Βρυξέλλες, τις μεταφέρετε στις πατρίδες σας, ε, στις χώρες σας, στις εταιρείες σας, στα πανεπιστήμια σας, γιατί ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα. Έχω πει πολλές φορές ότι η Ενεργειακή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει μόνο στις Βρυξέλλες, ε, με τις δικές σας τις προσπάθειες, στις πατρίδες σας, όχι μόνο διαδίδουμε αν θέλετε τα νέα, αλλά και αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπεται η οικονομία στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ πολύ και εκτιμώ ιδιαίτερα τι προσπάθειές σα και είναι χαρά και τιμή για μένα το να μπορώ να βρίσκομαι εδώ. Και έρχομαι πάντα όταν με καλείτε. Ο λόγο είναι ότι προετοιμάζεστε πάρα πολύ καλά για τι συζητήσει μα και οι συζητήσει σας είναι πάντα εύστοχε. Ε, έχουν ως στόχο να στηρίξουν τι κοινέ μα προσπάθειε ε, τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, την Επιτροπή και την Επιτροπή. Σα ευχαριστώ τον κύριο Κουλόν και τον κύριο Μπακ ε, για την πολύ σκληρή τους δουλειά που έκαναν για την ε, ανακοίνωση τη δική μας ε, σχετικά με έναν καθαρό πλανήτη για όλους. Έχετε δει το πόσο συμβατή είναι η σκέψη μας. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας και μπορούμε και να τα επικοινωνήσουμε αυτά καλύτερα στα κράτη-μέλη. Σήμερα λοιπόν συζητάμε ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει πάρα πολύ το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Ε, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες συνεδριάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως ξέρετε, σήμερα θα συζητηθεί κατά κύριο λόγο το κλίμα και τα ε, αξιώματα, το πώς θα επανδρωθούν τα αξιώματα. Τα δύο πάνε μαζί. Οι τελευταίες εκλογές κατέδειξαν με απόλυτη σαφήνεια ότι το θέμα του κλίματος κρίνεται επίγον θέμα από πολλούς ψηφοφόρους, κυρίως από τους νέους. Και επιτέλους στην Ευρώπη εξετάζουμε την κλιματική αλλαγή όχι μόνο ως κάτι το οποίο θα πρέπει να μας αναστατώνει και να μας κάνει να νιώθουμε μηχανία, αλλά και ως μια ευκαιρία που μπορεί να μας βοηθήσει να αναδιατάξουμε την οικονομία μας, να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο ζωής μας και επίσης ε, και να ε, δούμε το πώς πρέπει να οργανώσουμε τις οικονομικές μας δραστηριότητες. Ε, όλες λοιπόν τις ε, προκλήσεις που περιγράφω Όλα αυτά προσπαθούμε να τα συμπεριλάβουμε στη δουλειά μας ως Επιτροπή, να τα συμπεριλάβουμε στη μακροχρόνια στρατηγική μας που και αυτή θα συζητηθεί σήμερα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Όπως γνωρίζετε, τον Νοέμβριο του 2018 παρουσιάσαμε την ανακοίνωσή μας ε, με θέμα πώς μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη η οποία να μην ε, απειλείται από προβλήματα προβλήματα κλιματικής αλλαγής και παράλληλα να είναι και ευημερούσα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε θετική αντίδραση από τι επιχειρήσει από πολλού άμεσα ενδιαφερόμενου του οικονομικού τομέα Πολλοί είπαν ότι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν και αυτοί σε αυτή τη μετάβαση για κλιματική ουδετερότητα όπως αποκαλείται. Αυτά τα θέματα ε, παρουσιάστηκαν σε πολλές προεκλογικές εκστρατείες. Αυτό είναι το θέμα που όπως σας είπα συζητήσαμε ε, έντονα με τους πολίτες και κυρίως με τους νέους. Θέλω να πω, εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι αναλύσεις που κάνατε στις εκθέσεις σας ακολουθούν την κατεύθυνση το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και επίσης εσείς εστιάζεστε στο πώς η αλλαγή αυτή θα αλλάξει την ευρωπαϊκή οικονομία, τι θα σημαίνουν όλα αυτά για την ενεργειακή ασφάλεια και για τους πολίτες. Και όλοι καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξυγχρονίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως, πολλά εξαρτώνται από καλά προγράμματα, από την καλή θέληση, αλλά και το θέμα είναι πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά. Ένα κομμάτι αυτή τη έκθεση εστιάζεται σε εθνική, σε ενωσιακή χρηματοδότηση, στην ανάγκη να αλλάξουν οι επενδύσεις ε, και να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτείται η έρευνα και η καινοτομία. Αυτό που απασχολεί επίσης είναι πώς θα προσαρμοστούμε ε, κατά τις επόμενες δεκαετίες στις προκλήσεις του μέλλοντος. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί όλα αυτά τα χρειαζόμαστε για να ε, προσανατολιστούμε σωστά αν θέλουμε να επιδιώξουμε την κλιματική ουδετερότητα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ε, με αυτό που λέτε ότι η μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη. Δηλαδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε να βγάζουμε από το κάδρο τους πολίτες, τις περιφέρειες ή συγκεκριμένες ε, κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν μια δύσκολη φάση και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε αυτοί να μην ξεχαστούν. Γι' αυτό λοιπόν ε, μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση. Αυτό είναι το κλειδί, όχι μόνο για μας, αλλά και για την επόμενη Επιτροπή. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και την κοινωνική αποδοχή των προσπαθειών μας. Κρίσιμο αυτό για την επιτυχία μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η μετάβαση αυτή, τη μετάβαση αυτή θα πρέπει να την οικειοποιηθούν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Να προκύψει ένα είδος κοινωνικού συμβολέου ανάμεσα στις κυβερνήσεις, στις αρμόδιες αρχές, ε, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να εμπλακεί η κοινωνία και νομίζω ότι εδώ η Επιτροπή σας διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο γιατί εσείς είσαστε ο κρίκος που δένει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους πολίτες των κρατών μελών. Νομίζω ότι για την Επιτροπή σας ε, ε, θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να συμβάλλετε να προκαλέσετε εθνικές ε, περιφερειακές συζητήσεις ή συζητήσεις να είναι σωστά τεκμηριωμένες και να αφορούν όχι μόνο την θέσπιση της μακροχρόνιας ενωσιακής στρατηγικής, αλλά και το πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά και τι σημαίνουν για τις τοπικές κοινωνίες. Βεβαίως πρέπει να συνεργαστούμε με τους διεθνείς μας εταίρους. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει απομονωμένη σε αυτές τις προσπάθειές της, σε όλες τις συνεδριάσεις των G20, τον G7, στον ΩΣΑ. Η ε, Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει στην ε, προμετωπίδα, αλλά και όλοι οι άλλοι πρέπει να ακολουθήσουν. Ε, θα πρέπει αδιαμφισβήτητα να πρόκειται για ε, παγκόσμια προσπάθεια και όλοι να συμβάλλουν στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα διπλωματικά μέσα. Θα συμπεριλάβουμε την κλιματική αλλαγή ως, ένα, ως μια πολύ σημαντική παράμετρο για τις διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις μας. Ε, την κοινή αγορά, θα τη χρησιμοποιήσουμε ως κινητήρια δύναμη για την αλλαγή και θα επιμείνουμε στο σεβασμό του περιβάλλοντος ε, όταν ε, γίνονται εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω και πολύ λίγα λόγια για το δεύτερο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Είναι μια σύντομη έκθεση που αφορά στην τελευταία έκθεση για την κατάσταση ε, στην Ένωση περί ενέργειας, αυτή που εγκρίθηκε τον Απρίλιο. Έχουμε σημείωση πρόοδο στο να ε, υπάρχει πλέον ένα ε, αλληλένδετο ενεργειακό σύστημα στην Ευρώπη. Θα θυμάστε ότι το 2015 μιλάγαμε μόνο για ένα όραμα στρατηγικής και τότε υπήρχαν πάρα πολλές επιφυλάξεις για το τι μπορούμε να πετύχουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και τότε υποσχεθήκαμε ότι θα εφοδιάζουμε την Ευρώπη με ενέργεια που θα είναι ασφαλή, σε βιώσιμη, προσιτή και σήμερα νομίζω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όχι μόνο το πετύχαμε αυτό, αλλά πετύχαμε και πολλά περισσότερα. Από τότε που ξεκινήσαμε είχαμε αυτό που που πολλοί χαρακτηρίζουν ως μια βαθιά αλλαγή ε, των ενεργειακών μας συστημάτων, τη μεγαλύτερη από την δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Ανακαλύψαμε πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν βέβαια και σε άλλους τομείς. Και στο σημείο αυτό συζητάμε για αποκέντρωση, ε, για την απομάκρυνση του άνθρακα από την κατανάλωση. Μάθαμε το τι πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές έτσι ώστε να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και έτσι μάθαμε και το τι μπορούμε να κερδίσουμε αν χρησιμοποιήσουμε την ευφυή τεχνολογία. Όλα αυτά μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι στην Ευρώπη έχουμε όλα αυτά που χρειάζονται για να ε, υλοποιήσουμε το όραμά μας που είναι το 2050 μια Ευρώπη χωρίς άνθρακα. Χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι με τη βοήθειά σας εμείς στην Επιτροπή μπορέσαμε να υιοθετήσουμε όλες τις προτάσεις ε, που κατατέθηκαν για τη νέα στρατηγική, όλες αυτές που κατατέθηκαν και από το Κοινοβούλιο και από πολλούς άλλους. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη πλέον είναι σε θέση τη νέα δεκαετία να την ξεκινήσει με νέους κανόνες ε, οι οποίοι ε, θα είναι ε, εξυγχρονισμένοι και θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η κλιματική πρόκληση στον πλανήτη. Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης. Όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το ε, ποιος θα πρέπει να είναι ο πυρήνας της ε, Ενεργειακής Ένωσης, τότε οι περισσότεροι είχαν κατά νου την ενεργειακή ασφάλεια. Είχαμε λοιπόν τα ατυχήματα κατά το παρελθόν που γνωρίζετε. Είχαμε την ανακοπή ροής ε, εφοδιασμού αερίου σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Είχαμε ενεργειακές νησίδες όπως η χώρες της Βαλτικής, η Μάλτα και η Κύπρος, που δεν μπορούσαν να συνδεθούν με τους γείτονες, με τους εταίρους και έτσι βρισκόντουσαν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Σήμερα ε, είμαι στην ευτυχή θέση να σας πω ότι με την εξαίρεση της Μάλτας και της Κύπρου όλα τα άλλα κράτη-μέλη είναι σε θέση να προμηθεύονται αέριο τουλάχιστον από δύο διαφορετικές πηγές και το 2022 θα είναι τρεις αυτές οι πηγές αυτό ισχύει, όπως σας είπα, για όλα τα κράτη-μέλη, εξαιρουμένων των δύο νησιών μας γιατί δεν μπορέσαμε ακόμα να τα διασυνδέσουμε. Έχουμε όμως επενδύσει πάρα πολύ σε ε, τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου αερίου. Θεωρούμε ότι, μπας περιπτώσει, συνολικά είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για την ενεργειακή διασύνδεση και αυτό αφορά όχι μόνο τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες εξυγχρονίστηκαν με τα επιρροτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δουλέψαμε πολύ σκληρά και για να διασφαλίσουμε ότι οι γειτονές μας στα Βαλκάνια και αυτοί θα συνδέονται πολύ καλύτερα με ηλεκτρικό ρεύμα. Πιέζουμε να ε, βελτιωθεί η διασύνδεση, κάτι που στην περίπτωση τουλάχιστον των χώρων της Βαλτικής ήταν στο 0%. Τώρα είμαστε στο 20,3% γιατί υπάρχουν ε, οι διασυνδέσεις ε, στις χώρες της Βαλτικής, Σουηδία, Πολωνία και ε, σύντομα θα υπογράψουμε με τις χώρες αυτών των τριών κρατών ένα χάρτη πορείας που θα ολοκληρώσει τον εξυγχρονισμό με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα μέχρι το 2025. Γνωρίζετε ότι δουλεύουμε πολύ σκληρά για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε νέους στόχους 25% για το 2030 και για το στόχο αυτό πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό ως μια πρώτη προτεραιότητά μας γιατί αν πετύχουμε τους στόχο μας θα μειωθούν προφανώς ε, η, τα αέρια του θερμοκηπίου, θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια και θα βελτιωθεί η ποιότητα σε κτίρια όπου θα έχουμε καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Ένα από τα μαθήματα σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση, ένα που μάθαμε, είναι ότι όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα και ως εκ τούτου ε, πιο καθαρή κινητικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί με την παλιά τεχνολογία. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε, να κάνουμε μεγάλες επενδύσεις στα ηλεκτρικά οχήματα, στους νέους κινητήρες υδρογόνου και ε, εφόσον έχουμε να κάνουμε και με την ηλεκτρονική κινητικότητα, ήδη είμαστε πίσω. Ιδιαίτερα οι ανταγωνιστέ μας στην Ασία, ε, όπου έχουν αναπτύξει, μάλλον αναπτύσσουν αυτή τη τεχνολογία πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Γι' αυτό καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες για να δημιουργήσουμε αυτήν την, ε, την μπαταρία. Είναι η πολύ μεγάλη φιλοδοξία αυτή να, είμαστε, να γίνει αυτό το Airbus των μπαταριών. Έχουμε τώρα 160 εταιρείε που συνεργάζονται όταν, από τότε που φτιάξαμε αυτή την συμμαχία για την μπαταρία. Έχουμε 100 δις ε, επενδύσεις σε αυτό το project και τουλάχιστον τρία κονσόρτσια που συνεργάζονται. Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι το 2025 μέχρι το 2025 όταν δηλαδή η αγορά μόνο στην Ευρώπη θα είναι 250 δις για αυτές τις μπαταρίες μόνο στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να ηγηθούμε και να εξασφαλίσουμε ότι οι μπαταρίες που παράγονται στην Ευρώπη θα είναι ψηλή ποιότητα, πράσινες, βιώσιμες και θα έχουμε εγγύηση ότι και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο μέλλον θα είναι τα καλύτερα στον κόσμο και από την άποψη του μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα. Με όλες αυτές τις προσπάθειες που σας περιγράφω και με όλους αυτούς τους στόχους που έχουν ε, ε, εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μέχρι το 2030 υπολογίζουμε ότι θα έχουμε περικόψει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 40%. Εάν ε, υλοποιηθούν όλα μας τα ενεργειακά προγράμματα θα φτάσουμε το 45% μείωσης και έτσι θα αποδείξουμε αυτό που ήταν τόσο σημαντικό και που εξέπληξε τόσο κόσμο όταν γίνονταν οι διαπραγματεύσει στο Παρίσι να θα αποδείξουμε ότι μπορούμε μια τόσο μεγάλη οικονομία να περιορίσει τους, ε, τις εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου κατά 22% και να αναπτύξεις την οικονομία σου ε, ταυτόχρονα. Εάν εξισορροπήσουμε σωστά τα πράγματα, έχουμε, ε, έχεις αποτελέσματα. 1,4 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης είναι στον τομέα της ενέργειας από αυτές που δημιουργήθηκαν το τελευταίο καιρό και τα νούμερα αυτά θα αυξηθούν κι άλλο ε, κανονικά. Και να κλείσω με ένα άλλο θέμα από το οποίο συζητήσαμε τον κύριο Κούλον, όταν, καθώς ερχόμασταν εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Ε, πρόκειται για την ε, αποδοχή και για το έμφαση στον κόσμο, ε, στους πολίτες και τη σημαντική επικοινωνία με τις περιφέρειες που περνούν δύσκολες φάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις και σε όλες τις χώρες όπου έχουμε φτωχότερες περιφέρειες ε, έχουμε τέτοιου προ... τέτοια προβλήματα και γι' αυτό και η δημιουργία μιας πλατφόρμας για ε, τις περιφέρειες που χρησιμοποιούν περισσότερο άνθρακα ήταν σημαντική. και αυτό βλέπουμε εκεί μαζί τι κάνουμε, αν πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αν πρέπει να αυξήσουμε περισσότερο τις προσπάθειες, ώστε κάθε μια από αυτές τις περιφέρειες να μπορέσει να αποκτήσει μια νέα προοπτική, ε, τόσο για τον άνθρακα όσο και για την οικονομία. Και ο καθένας που εργάζεται σε αυτές τις περιφέρειες να έχει εγγύσεις για καλύτερη ζωή και καλύτερες ποιότητες ε, απασχόληση. Η συνεργασία δεν είναι εξαιρετική. Το πρόγραμμα που έχουμε προτείνει για να συνεργαστούμε με αυτές τις περιφέρειες που θέλουν να δουλέψουν μαζί μας ε, ε, δουλεύουμε για νέα οικονομικά project για το μέλλον. Αφήνουμε τις περιφερειακές αρχές να διαλέξουν τα project πιστεύουν πως, που πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν και ψάχνουμε και τα χρήματα μαζί. Είτε πρόκειται για αναδιανομή μέσω του Ευρωπαϊκού ε, Επενδυτικού Ταμείου ή άλλων ε, χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ε, την κάθε περιφέρεια που θέλει να αναπτύξει νέα οικονομικά μοντέλα. Και αυτή θα είναι προτεραιότητα και για την επόμενη Επιτροπή, την επόμενο Κοινοβούλιο, γιατί μιλάμε για 200.000 ανθρακορίχους αλλά και για πάρα πολύ κόσμο ακόμα που έμεσα ή άμεσα απασχολείται στον τομέα του άνθρακα. Να πω και κάτι και για την ενεργειακή φτώχεια. Έχουμε κάνει πολλά, αλλά ακόμα 50 εκατομμύρια κόσμο στην Ευρώπη έχει πρόβλημα να πληρώσει το λογαριασμό ενέργειά του στο τέλο του μήνα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη πω όλε αυτέ οι μεταρρυθμίσει που ξεκινάμε και που εφαρμόζουμε θα πρέπει να έχουν και αυτό αυτή την πολύ σημαντική κοινωνική πτυχή υπόψη, ώστε ο κόσμος να το δεχτεί ως μια δίκαιη προσέγγιση που τελικά βελτιώνει την ποιότητα της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς όλα τα κράτη-μέλη ε, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες αναλύσεις όσον αφορά τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια ε, τα έχουμε λάβει από όλες τις χώρες μέλη και θα τα ε, τελειοποιήσουμε σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και πιστεύω πως αυτό το τελευταίο κομμάτι του παζλ θα εξασφαλίσει πως η Ενεργειακή Ένωση δεν θα είναι μόνο πλαισιωμένη, δεν θα καλύπτεται μόνο από την νομοθεσία αλλά θα εφαρμόζεται όλα σε επιτόπου και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ζητήσω τη βοήθειά σας γιατί εσείς είστε οι πρεσβευτές μας στα κράτη-μέλη. Ε, εσείς πρέπει να μιλήσετε για αυτά τα θέματα, να θέσετε τις σωστές ερωτήσεις και να εξασφαλίσετε πως όλη η δουλειά που κάνουμε εδώ θα εφαρμοστεί και θα υλοποιηθεί στα κράτη-μέλη μας. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και που δημιουργήσατε αυτή την ευκαιρία ώστε να σας παρουσιάσω τα πορίσματα της κοινή μας προσπάθειας τα τελευταία πέντε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αν κάποιος είχε κάποια αμφιβολία, να άλλη μια απόδειξη για το πόσο σημαντικό είναι το έργο που έχει επιτελεστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και τους τελευταίους μήνες, γιατί αναφερθήκατε στην ε, Ενεργειακή Ένωση. Τώρα θα δώσουμε το λόγο πρώτα στον Πιέρ Ζαν Κουλό και τον Στέφαν Μπακ που είναι οι συνεισηγητές στο θέμα της στρατηγικής αυτής. Άλλο ο Σκουλών και ο πρόεδρος ε, του τμήματός μας. Οπότε, πέντε λεπτό καθένας παρακαλώ. Πρώτος, ο Πιεριζό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την πρόεδρε Σεύκοβιτς. Ε, συνεργαζόμαστε εδώ και πέντε χρόνια πάρα πολύ καλά και όταν λέω συνεργαζόμαστε, το εννοώ. Γιατί αν ε, σήμερα παρουσιάζουμε κάποιες σκέψεις όσον αφορά την μακροπρόθεσμη στρατηγική για μια ευημερούσα οικονομία, σύγχρονη, ανταγωνιστική και ουδέτερη όσον αφορά το κλίμα, πρόκειται για ένα επίτευγμα, αλλά πρόκειται και για ένα σημείο κίνησης. Επίτευγμα μετά από μια διαδικασία συνεχών διαβουλεύσεων ανάμεσα στην ΟΚΕ και το τμήμα του οποίου εγώ προεδρεύω, ε, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς, αλλά επίσης και με τον Επίτροπο Άρια κανιέτε και με τις υπηρεσίες των διάφορων γενικών διευθύνσεων. Διότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει υποχρεωτικά μια συνεργασία για να πετύχουμε το έργο μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε αντιπαράθεση ή να ξεχάσουμε τις μεταφορές και να πούμε ότι είναι λιγότερο σημαντικές από την ενέργεια ή να παραβλέψουμε τις μεταφορές και την ενέργεια όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι για το περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουμε τον πολίτη ε, και να αφήσουμε μόνο τους πολιτικούς να αποφασίζουν ή να βάλουμε στην πάντα τα συνδικάτα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, είναι μια υποχρέωση που έχουμε να συνεργαζόμαστε επιμονή μου βάσεως, να έχουμε επιμονή μου βάσεως διάλογο. Και είναι κάτι υποχρεωτικό σε αυτό το τομέα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονών μας και όχι τόσο του πλανήτη όπως συνεχίζουμε να λέμε γιατί ο πλανήτης έχει νόημα όταν ε, βοηθάμε αυτούς οι οποίοι ζουν πάνω σε αυτό το πλανήτη. Χρειάζονται λοιπόν προσπάθειες και εδώ και χρόνια χάρη στο έργο ε, της Επιτροπής ε, το συνεχές, το μόνιμο και βλέπω εδώ στην αίθουσα τους συνεργάτες του Αντιπροέδρου με τους οποίους συνεργάτες έχουμε επαφές ε, τακτικότατα. Βλέπω και τα μέλη της γραμματείας του τμήματός μας οι οποίοι επίση συνεργάζονται με τους διάφορους εκπροσώπους εδώ. Υπάρχει μια συνεχή συνεργασία ε, υπέρ του πολίτη, για το μέλλον του πολίτη, γιατί αυτό το μέλλον είναι σήμερα, όπως μας λέει ο Επίτροπος, για να μην πούμε ότι ήταν χτες. Θυμάμαι ότι αποτελούσα μέρος των αντιπροσωπιών στο Μπουρζέ. Ε, συνεργαζόμαστε για αυτό το θέμα ήδη και έχουμε υπογράψει όλοι μαζί μια ωραία συμφωνία, η οποία πρέπει όμως να γίνει και πράξη. Και τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει πραγματικά να συμμετέχουν. Και σήμερα θέλω να σας εκφράσω την ανησυχία μου, αγαπητοί συνάδελφοι. Και αυτό διότι βλέπω επιχειρήσεις, και το λέω ξεκάθαρα, πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλές, την πλειοψηφία, που τι κάνουν, τους ενδιαφέρει το έργο αυτό και προσπαθούν και τη συγχαίρω. Βλέπω και τους πολίτες που και αυτοί αναλαμβάνουν το δικό τους το κομμάτι. Η Συνομοσποδία εργατών, για παράδειγμα, πρόσφατα υπογράμμισε αυτό το ζήτημα. Όμως, συγχρόνως, βλέπω κάποιες χώρες μέλη να σέρνουν τα πόδια, να καθυστερούν. Όταν τα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα αρχίζουν να παίρνουν μορφή και τα έχουμε συζητήσει πολύ με τον Αντιπρόεδρο Σεφκοβιτς, πολύ φιλικά, για κάποιες χώρες δυστυχώς, ακόμη και στη χώρα εδώ στην οποία βρισκόμαστε, είναι σε καταστροφική κατάσταση. Αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουμε, έχουμε υποχρέωση με όλους τους συμμετέχοντες, όλοι μαζί που εκπροσούμε τις επιχειρήσεις, όλοι μαζί που εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών, την οργανωμένη, την πλήρη σύνθεσή της, όλοι εμείς που εκπροσωπούμε ε, συνδικάτα και εργαζόμενους στις χώρες μας, έχουμε την υποχρέωση να πιέσουμε, να ανασκουμποθούμε και να πιέσουμε, πολύ να πιέσουμε τους πολιτικούς της χώρας μας, ώστε να αντιληφθούν τι είναι αυτό που είναι αναγκαίο και τι σημαίνει αυτό που υπέγραψαν πριν από λίγα χρόνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, μας μένει πολλή δουλειά και θα την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και όταν έχουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάμε να τους δούμε και αυτή τη γνωμοδότηση που θα ψηφίσουμε θα το την πάμε. Θα την πάμε στο νέο επίτροπο που θα είναι αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα. Θα την πάμε και θα την εξηγήσουμε στους προέδρους ε, των διαφόρων οργάνων και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα είναι αρμόδια για αυτό το θέμα. Θα το κάνουμε. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που ακούσαμε. Στέφαν Μπακ τώρα. Ε, θα ακούσουμε τη δικιά σας την πλευρά με τον ίδιο ενθουσιασμό, ε? στα Σουηδικά αυτή τη φορά. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο για τη δουλειά που έχει κάνει για την ανακοίνωση αυτή. Ε, πραγματικά προσβλέπουμε στο να έχουμε μια συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μας για τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα. Εμείς ε, προσβλέπουμε ε, στο να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Θέλουμε να υπάρχει μια ουδέτερη κλιματικά οικονομία. Ε, επίσης στηρίζουμε τις προτεραιότητες που αναφέρονται στην έκθεση της Επιτροπής. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ποια είναι τα μέτρα τα οποία εμείς κρίνουμε απαραίτητα για να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο για το κλίμα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν χρειαζόμαστε μια γρήγορη στρατηγική για την περίοδο 30, 2030 έως 2050. Αυτό πρέπει να το έχουμε έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε στις αποφάσεις ε, που έχουν ληφθεί. Πολλές εξ αυτών θεωρούν ότι το 2030 είναι η καταληκτική ημερομηνία. Εμείς ε, έχουμε πολλές γνωμοδοτήσεις όπου γίνεται λόγος για την κυκλική οικονομία, την ψηφιοποίηση, την ε, συμμετοχική οικονομία. Όλα αυτά ε, μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων ε, με ε, μικρότερες εκπομπές. Η προβλεψιμότητα, ο προγραμματισμός, αυτά είναι θέματα που πρέπει να διασφαλιστούν και όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας προς τις τρίτες χώρες, και την ε, κλιματική αλλαγή, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει μια συμμαχία για μετάβαση, να υπάρχουν ε, ήδη και ίσοι όροι για τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσον αφορά στον ανταγωνισμό. Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο να αποδείξει ότι η απαραίτητη μετάβαση θα αποβεί θετικά για το σύνολο της κοινωνίας. Εξάλλου στηρίζουμε την άποψη ότι όλοι οι ενεργειακοί πόροι που δεν έχουν σχέση με την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, όλοι αυτοί οι πόροι θα πρέπει να την χάνουν καλύτερη εκμετάλλευση, ε, να υπάρχει ευελιξία. Η βιοενέργεια είναι πολύ σημαντική, όπως ε, και οι καταβόχτρες διοξιδίου του, φυσικές διοξιδίου του άνθρακα. Η κινητικότητα είναι απαραίτητη για την ε, εύρυθμη λειτουργία της κοινή αγοράς ε, και πρέπει να περιορίσουμε την, ε, το αποτύπωμα άνθρακα στην κινητικότητα, η οποία μας είναι σημαντική και πρέπει και αυτή, και αυτή να περασπιστούμε. Η χρηματοδότηση των μέτρων είναι απαραίτητη για να έχουμε προγράμματα επίδειξης, να έχουμε νέες πρωτοβουλίες, ε, να κινητοποιηθούν οι δημόσιοι πόροι, έτσι ώστε να μπορούμε και να κινητοποιήσουμε πράσινες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Επίτροπε, εσείς ε, αναφερθήκατε επίσης σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό είναι κάτι που όλοι μας στηρίζουμε κατά τη μεταβατική περίοδο. Τα κρατημέλη, οι περιφέρειες, οι τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι ε, στην αγορά εργασίας και το υπόλοιπο της κοινωνίας των πολιτών όλοι πρέπει να συμπεριληφθούν. Η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει εις βάρος ε, κάποιων ομάδων ε, της κοινωνίας, γιατί αλλιώς θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα. Έχουμε και μία πρόταση που αφορά στην ε, κλιματική αλλαγή, ε, μία επιτροπή θα κάνει επιστημονικές αναλύσεις και μετά θα καταθέσει προτάσεις. Καλούμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να συστήσουν τις δικές τους τις επιτροπές εκεί όπου δεν τις έχουν και θεωρούμε επίσης ότι είναι επιγόντως απαραίτητο να έχουμε διάλογο με τους πολίτες ε, για να γίνουν αποδεκτά τα μέτρα που εμείς κρίνουμε απαραίτητα ε, κατά τα επόμενα χρόνια που θα προσπαθήσουμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας. Θα πρέπει ε, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε εθνικό, περιφερειακό, οποιοδήποτε άλλο επίπεδο να είναι απαραίτητος, να προηγείται απαραίτητα ο διάλογος. Εμείς ήδη συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και θέλουμε να συμμετέχουμε και στο μέλλον. Η ε, συνέχιση της ε, μετάβασης, η διεύρυνση της βάσης, αυτά είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ και για το πάθος με το οποίο μιλήσατε στα Σουηδικά. Και τώρα λοιπόν μπαίνουμε στη συζήτηση με τα μέλη ε, και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας να μην ξεπεράσετε ε, το χρόνο που προβλέπετε για να παρέμβετε γιατί ο κύριος Επίτροπος έχει και άλλες υποχρώσεις. Για τα κάτσο παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, εκ μέρου των εργοδοτών, Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, σας καλωσορίζουμε και εμείς και πολύ σύντομα θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και οι κλάδοι εκείνοι που χρησιμοποιούν πολύ εντατικά την ενέργεια θέλουν να προχωρήσουμε και να πετύχουμε τους στόχους των Παρισίων. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή λύσεων χαμηλού άνθρακα. Για να πετύχουμε όμως τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κλιματική στρατηγική, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για την μετάβαση αυτή. Πολύ σύντομα λοιπόν. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης για να αναπτύξουμε τέτοιες τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα. Χρειαζόμαστε επίσης πολιτικά μέτρα για να διατηρήσουμε την παραγωγή χαμηλού άνθρακα τόσο στις εσωτερικές μας αγορές όσο και πιο έξω. Και έπειτα χρειάζεται και πρόσβαση σε ενέργεια χαμηλού άνθρακα με ανταγωνιστικό όμω. κόστος. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή για την απάλληψη του άνθρακα, αλλά θα πρέπει να πιέσει και άλλους εταίρους να επιδείξουν την ίδια φιλοδοξία μέσω διπλωματικών προσπαθειών. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τους δύο συγητές για το εξαιρετικό τους έργο. Ευχαριστούμε. Γιάτσεκ. Όλιβερ Ρέπκε τώρα, Αυστρία. Τμήμα 2. Ε, εκ μέρους των εργαζομένων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όντω, εκ μέρου των εργαζομένων, Αντιπρόεδρε, καλώ ήρθατε στην ΟΚΕ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σα έχουμε μαζί μα σήμερα και ξέρουμε πω έχετε αναλάβει την δέσμευση να προωθήσετε τον διάλογο, τον κοινωνικό διάλογο, τον διάλογο με του κοινωνικού εταίρου. Κάθε φορά χαίρομαι όταν βρισκόμαστε μαζί σα, τα συνδικάτα, οι κοινωνικοί εταίροι. Και αυτό είναι ένα λόγο για τον οποίο ελπίζουμε να παραμείνετε επίτροπο και στην επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, ως ομάδα των εργαζομένων, τα δικαιώματα και μια δίκαια μετάβαση είναι στοιχεία κλειδί για μας. Οπότε, όταν διαβάσουμε το πρώτο σχέδιο του Συμβουλίου, οι στρατηγικοί στόχοι δηλαδή που θα εγκριθούν αύριο, ανησυχήσαμε και απογοητευτήκαμε κάπως. Ε, τα θέματα της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων μόλις μεταβίας αναφέρονται στο κείμενο. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω και να παραβλέψουμε τα επιτεύγματα της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όταν πρόκειται για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, η πρόκληση θα είναι να ξεπεράσουμε κάποια συμφέροντα και να καταφέρουμε να πετύχουμε μια κοινωνική συνένεση. Οι πολίτες θέλουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτήν την ε, άμεση πρόκληση και να λάβουμε υπόψη μας τις συνέπειες των πολιτικών για το κλίμα, προκειμένου η στρατηγική για το κλίμα να είναι επιτυχής. Και θα ολοκληρώσω υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα μου, όπου εκπροσωπούνται πάνω από 80 συνδικαλιστικές οργανώσεις, θέλει να στείλει ένα σαφές ε, μήνυμα στα μέλη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων της θετίας αυτής για να ε, διασφαλίσουμε αυτό που είπατε και εσείς πριν, να μην μείνει κανείς πίσω σε αυτήν την τεράστια διαδικασία αλλαγών, σε αυτήν την μετάβαση. Κανένας, κανένας κλάδος, κανένας τομέας, καμία κοινότητα, καμία περιφέρεια, κανένας πολίτης. Είναι στοιχείο κλειδί αυτό αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την άνοδο του λαϊκισμού και του εξτρεμισμού που τρέφεται από το αίσθημα αδικίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε σήμερα και προσβλέπουμε στην μελλοντική συνεργασία μας ε, μαζί σας, ελπίζοντας να παραμείνετε επίτροπος. Ευχαριστούμε, Όλιβερ. Κάρλος Τρίας Πίντο, τώρα, από την ομάδα 3. Ευχαριστώ, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ, Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε. Πριν από 10 χρόνια εδώ στην ΟΚΕ, παρουσίασα μια έκθεση πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επένδυση. Και πέρυσι ήμουν εισηγητής προγράμματος δράσης της Επιτροπής μας για την βιώσιμη ανάπτυξη και τα βιώσιμα, τις βιώσιμες επενδύσεις. Κάτι το οποίο σήμερα ε, βρίσκει ε, τη διαμόρφωσή του μέσα στο Invest EU. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε βιώσιμα ε, οικονομικά και βιώσιμες επενδύσεις στη νέα αυτή οικονομία, την βιώσιμη, με συγκεκριμένα κριτήρια. Όπως έκανα και εγώ στην ε, ΟΚΕ, ε, πρέπει και εσείς να υπογραμμίσετε ότι χρειαζόμαστε στοιχεία αξιόπιστα και συγκρίσιμα μεταξύ τους, όχι μόνο για τις επιπτώσεις που έχουν επενδύσει αυτές πάνω στο κλίμα, αλλά χρησιμοποιώντας διάφορους ε, διάφορα κριτήρια και περιβαλλοντικά και κοινωνικά και διακυβέρνησης. Είναι κάτι το οποίο συνάδει και με το κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο. Και ευθυγραμμίζεται και με τις δικές μας εκθέσεις Και ολοκληρώνω. Συγχαίρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητούμε να συνεχιστεί αυτή η δέσμευση υπέρ της βιωσιμότητας. Ευχαριστούμε. Ο συνεχίζουμε Είπαμε να τηρείτε το χρόνο σας. Ούντο Έμερλινγκ τώρα. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εδώ βρίσκομαι. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για το όραμα του 2050 για να έχουμε μια οικονομία ουδέτερη σε επίπεδο κλίματος. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ότι όταν μιλάμε για τους στόχους του 2030. Στόχοι δηλαδή οι οποίοι συζητήθηκαν από αυτήν την Επιτροπή και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και θεωρώ ότι αυτούς τους στόχους ε, για το 2030 μπορούμε να τους επιτύχουμε στα κράτη-μέλη και αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος Κουλόν το είπε ότι βέβαια πολλά κράτη-μέλη ε, δυσκολεύονται αυτούς τους στόχους να τους υλοποιήσουν με συγκεκριμένα μέτρα και επιτρέψτε μου εδώ να αναφερθώ στο θέμα του διοξιδίου του άνθρακα. Εγώ θεωρώ ότι ε, έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα για την οικονομία, για τους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να αναπροσανατολιστούν προς ε, την κατεύθυνση ε, του να υπάρχει μια οικονομία χωρίς ε, άνθρακα και χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι η διατροφή. Στη Συμφωνία των Παρισίων ε, προβλέπεται ιδιαίτερος ρόλος ε, για τα θέματα ε, διατροφής, γεωργίας, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το θέμα διατροφή ή και τρόφιμα αν θέλετε είναι η προϋπόθεση για όλα τα άλλα. Η εξασφάλιση των τροφίμων είναι συνεκουανών. Έχουμε βεβαίως το παρεπόμενο, την εκπομπή ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στη Γεωργία θα μπορούσαμε να καταφύγουμε σε άλλα όμως ε, μέτρα να έχουμε πιο αποτελεσματική οικονομία να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας αλλά κυρίως ε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιοενέργεια και τη δέσμευση του άνθρακα και στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω την έκθεση του συναντέλφου που μιλάει για τη δέσμευση του άνθρακα μέσα από τη φωτοσύνθεση Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Εμίλ Μάκινα από τη Σλοβακία. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής και εύχομαι καλή επιτυχία και για το μέλλον. Ποιότητα της ζωής τώρα δεν εξαρτάται από την αύξηση του ΑΕΠΑ αλλά περισσότερο από το περιβάλλον ε, στο οποίο μέσα ζούμε. Και αυτό είναι πρόκληση όχι μόνο για τους πολιτικούς, αλλά και για την κοινωνία των πολιτών. Σήμερα οι πολιτικοί συνήθως ε, βάζουν βραχυπρόθεσμους στόχους, γιατί αυτό έχει πιο μεγάλο πολιτικό αντίκτυπο όμως ε, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, ε, όπως το περιβάλλον, είναι ε, πιο δύσκολο να πείσουν τον κόσμο ότι είναι πιο σημαντικοί. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας θα πρέπει να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες, να επενδύσουμε άρα περισσότερο στην επιστήμη και στην τεχνολογία και από κοινού να δούμε τι θα προωθήσει ε, ε, την ποιότητα αυτή της ζωής που θέλουμε. Είμαι βέβαιος ε, ότι μπορούμε αυτά να τα πετύχουμε οι στόχοι είναι σαφείς και εξαρτάται από μας να ε, δώσουμε τη σωστή εικόνα, να δώσουμε τη σωστή ενημέρωση στον κόσμο και να επιτύχουμε τους στόχους που επιθυμούμε. Ε, θέλω λοιπόν να στηρίξω όλους όσοι θα συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες ή μάλλον συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες στις χώρες μας. Ε, ελπίζω πως η εργοδότες και οι, απασχο... και οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να συμμετέχουν ε, στην επιτεύξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ, Εμίλ. η κυρία Μιλτόβιτς από την Λετωνία. Ευχαριστώ. αγαπητέ κύριε Σεύκοβιτς, πραγματικά εκτιμώ τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Θα ήθελα να, να στρέψω την προσοχή σας στο γεγονός ότι μαζί με τους συναδέλφους εργαζόμαστε για την επικοινωνία και για την πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Σημαντικό έγγραφο είναι αυτό γιατί προτείνουμε πλαίσιο για την ενέργεια και ε, ε, Επίσης, τη μετακίνηση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία για τα θέματα τον του ενεργειακού φόρου. Οι, οι πρωτοβουλίες για τον φόρο στην ενέργεια είναι οι πιο σημαντικές, πιστεύουμε, γιατί ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τις κλιματικές αλλαγές. Θα ήθελα επίσης να στρέψω την προσοχή σας στο ότι τα κοινωνικά θέματα θα πρέπει να είναι ε, μια από τις προτεραιότητες. Να σας θυμίσω ότι η Η ισότητα ε, ε, των εισοδημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, θα πρέπει να επιτευχθεί και υπάρχει κόστος λόγω της ενεργειακής μετάβασης όσον αφορά την ψηφιοποίηση της ενέργειας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ λοιπόν προσεκτικοί όσον αφορά την φορολόγηση των, της ενέργειας. Λοιπόν, για το σύστημα συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα είναι ευπρόσδεκτο, αλλά ε, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στηρίζοντα τον διάλογο και θα πρέπει να συμμετέχει σε συζητήσεις. Αναφέρατε επίσης ε, την ε, δικαιοσύνη στην μετάβαση και μεταναφερθήκατε και στην ενεργειακή φτώχεια που όντως υπάρχει και μάλιστα αυξάνεται από το κίνημα των καταναλωτών ε, στην Ευρώπη θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να σκεφτείτε και να προτείνετε πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε κοινού ορισμούς ε, για την ενεργειακή φτώχεια και που θα καλύπτουν όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο θα μπορέσει να μας κάνει να προχωρήσουμε με αυτές τις πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ε, κοινοτήτων, δήμων και κοινοτήτων. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Η κυρία Ζέρμινα Ντουμπράφσκα τώρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σεύκοβιτς και ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Είμαστε ευτυχείς που ήρθατε σε αυτή τη συνεδρίαση κύριε Σεύκοβιτς. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ασχοληθούμε με τον μέλλον ήδη από τώρα. Πρέπει να βρούμε κοινέ προσεγγίσεις. Όμως αυτές οι κοινέ προσεγγίσεις θα πρέπει να ε, αξιολογούνται ε, το ίδιο για όλους. Καθαρός πλανήτης για όλους σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε και να το πετύχουμε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλοι πρέπει να προσπαθήσουν να πετύχουν αυτό το στόχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει το 10% μόνο των παγκοσμίων εκπομπών. Το υπόλοιπο 90% παράγεται αλλού. Εμείς έχουμε βάλει φιλόδοξους στόχους που είμαι βεβαία ότι θα καταφέρουμε να τους επιτύχουμε, όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, ότι είναι και δίκαιοι ε, ε, εντός της Ένωσης. Εντός της Ένωσης πρέπει να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά, αλλά να μην ξεχνάμε ότι επίσης εντός της Ένωσης πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και όχι να αποδυναμωθούμε. Και το λέω αυτό γιατί, γιατί η γεωργία, που είναι ένας τομέας που εγώ εκπροσωπώ, οι απαιτήσει έχουν ε, οριστεί από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε να εισάγονται υπηρεσίες και αγαθά που παράγονται αλλού και υποτελείως διαφορετικές συνθήκες. Ε, γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ζητήσω να σκεφτείτε τους Ευρωπαίους γεωργούς και να προσπαθήσετε εξ ονόματός τους να επιμείνετε ώστε οι απαιτήσει να είναι οι ίδιες. Σε όλες μας λοιπόν τις διαπραγματεύσεις να ε, ε, μιλάμε και για υποχρεώσει τη άλλη πλευρά. Γιατί διαφορετικά αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον μα και εναντίον των Ευρωπαίων πολιτών. Σα ευχαριστώ και πάλι και θα ήθελα να σα ευχηθώ καλή επιτυχία για την επόμενη ε, θητεία. Και επίση εύχομαι να λάβετε πολλές και σοφές ε, αποφάσεις. Φορμαία τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Σεφτοβίτς, μεγάλη τιμή για μας και πολύ χαίρομαι που αναφερθήκατε σε όλες μας τις ανησυχίες στην ε, αρχική σας ε, εισήγηση που έχει να κάνει με τον άνθρακα, με τις εξορίξεις τις διάφορες περιφέρειες κτλ. Η πλατφόρμα η οποία λειτουργεί είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τις περιοχές που έχουν εξορίξεις και θα συνεχίσουμε το έργο μας. Όμως τι λένε Τώρα, φάκτα non verba. Γιατί το λέω αυτό επειδή ο πρόεδρος μας έρχεται από την Ιταλία. Οπότε, πρέπει δηλαδή να υπάρχει αντιστοιχεία λόγων και πράξεων. Η Επιτροπή των Περιφερειών, ο κύριος Λάμπερτς, είπε ότι οι χώρες μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από το 21 μέχρι το 27 θα πρέπει να αφιερώσουν προπολογισμό για να συνοδεύσουν στις εξορρυκτικές περιφέρειες την ενεργειακή μετάβαση. Θα ήθελα λοιπόν σχόλια από εσά και να μας πείτε αν θα ακολουθήσετε αυτή την πρόταση στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Όντω, οι πράξεις πρέπει να ακολουθούν τα λόγια, να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στα δύο. Ναι, βεβαίω, Ιρλανδία τώρα. Μπόλαντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Σας καλωσορίζω κι εγώ εδώ και σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε που αναφερθήκατε στη δικαιοσύνη και στην δίκαια μετάβαση που αναγνωρίζετε ότι είναι πολύ βασικό αυτό. Ελπίζω να συνεχίσετε να βασίζεστε σε αυτό, σε όλη την ενεργειακή μετάβαση. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέρφους που τους συνεισηγητές δηλαδή όταν μίλησαν για την διαβούλευση γιατί πράγματι ένα από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή μετάβαση είναι ακριβώς η φορολόγηση χωρίς προηγουμένως να έχουν υπάρξει διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. Με η φορολόγηση είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους και τους οδηγεί στη φτώχεια συχνά. Αν λοιπόν έχετε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη μετάβαση, ε, δεν πρέπει να τους κατηγορείτε για λαϊκισμό ή επειδή ψηφίζουν ακραία κινήματα συμφωνούν με αυτά όχι επειδή τους αρέσουν, τα αγαπούν κτλ, αλλά γιατί είναι τα μόνα κινήματα τα οποία εκφράζουν τους φόβους τους. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας λοιπόν και να, να βασίσουμε τη στρατηγική μας στην δικαιοσύνη. Επίσης θέλω να πω ότι όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές, κυρίως τις μεταφορές, και κυρίως στις αγροτικές περιοχές, στην Ήπεθρο, να ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα και ότι προσθέτει κόστος στις οικογένειες που ζουν στην Ήπεθρο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το θέμα αυτό των μεταφορών το αντιμετωπίζουμε παρκώς στην στρατηγική αυτή. Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Τέλος, κάθε χώρα χρειάζεται τη δικιά της διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή. Σκεφτείτε το αυτό σαν τμήμα της πολιτικής σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάντως για το έργο σας και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Αλμπέρτο Ματσόλα τώρα, Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εγώ θα μιλήσω Ιταλικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μου ως Επιτροπή ε, συμμεριζόμαστε αυτή τη στρατηγική που παρουσιάστηκε και όλες αυτές τις εργασίες που έχουν γίνει για το, την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2050. Όμως, θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στο θέμα της ενέργειας ε, που είσαστε αρμόδιος, ε, προβλέπετε ανανέωση όλου του, όλης της παραγωγής και αυτό για να είμαστε εξυγχρονισμένοι, να έχουμε έχουμε μια οικονομία χωρί τη χρήση άνθρωκα. Αλλά δηλαδή πρέπει να γίνουν μεγάλε προσπάθειε, κυρίω στο θέμα το ψηφιακό. Για τι ε, μεταφορέ, ε, εκεί πράγματι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιοποίηση, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουμε και μια ουσιαστική μετάβαση. Τώρα, φτάνω σε κάποια προβλήματα. Έπεα που αναφέρει ένα λατινικό ρητό ότι ε, επεαπτερώντα, αλλά οι πράξεις παραμένουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιες είναι οι απαραίτητες επενδύσεις. Στον τομέα της ενέργειας έχουμε κάθε χρόνο 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ε, στις μεταφορές 9 δις. Για να μην μιλήσουμε για την ε, θέρμανση στις κατοικίες για να μην υπάρχει χρήση του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι για περίπου 30 χρόνια θα πρέπει δύο μήνες το χρόνο να ε, παρεμβαίνουμε για να μπορούμε να στηρίξουμε αυτές τις επενδύσεις. Αυτό μπορεί να γίνει. Πάρα πολλοί μίλησαν για το κατά πόσο αυτό είναι αποδεκτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Και η αποζημίωση αυτών των επενδύσεων σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια εξοικονόμηση ενέργειας ε, τη τάξη του 50%. Και δύο ερωτήσεις. Πώς μπορούμε αυτή τη στρατηγική να την παρουσιάσουμε ε, στους πολίτες ε, χωρίς να υπάρχουν αρνητικές παρενέργειες. Πού θα βρούμε αυτά τα χρήματα που είναι απαραίτητα. Θα χρειαζόταν ίσως 15 φορές ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότηση όπως αυτό του κυρίου Γιούγκερ, στρατηγικών επενδύσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η κυρία Μαρία Μαγέροβα από τη Σλοβακία. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνετε, ε, όχι μόνο ως μέλος της ομάδας των εργαζομένων, αλλά και ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου, η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τον κόσμο και πλέον ε, υπάρχει αστάθεια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, σε αυτή την κατεύθυνση. Ο στόχος όλων μας είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι πολύ σημαντικές σε επίπεδο στρατηγικής. Αυτές οι διαβουλεύσεις έλαβαν χώρα σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι ομάδες στόχοι ήταν επαγγελματικοί φορείς, ομάδες πολιτών, ε, περιφερειακές και τοπικές αρχές και βεβαίως και οι πολίτες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, σε αυτή την κατεύθυνση μια ε, αλλαγή της οικονομίας μας προς την κατεύθυνση των μηδενικών εκπομπών θερμοκηπίου. Αυτό απαιτεί να ε, δοθούν στους πολίτες οι απαραίτητες πληροφορίες, να τους ενημερώσουμε ότι αυτή η αλλαγή είναι πραγματικά αναπόφευκτη. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη για το μέλλον. Και τέλος από τη Φινλανδία ο κύριος Τάινεμ για δύο λεπτά. Τάινεμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω φινλανδικά. Αξιότιμε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που έρχεστε και πάλι εδώ για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ έρχομαι από τη Φινλανδία και εκπροσωπώ τους ε, γεωργούς ε, και ιδιοκτήτες δασών της ε, Φινλανδίας. Και γι' αυτό θέλω να δείξω ένα θέμα που αφορά στο δυναμικό που έχει η βιοοικονομία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι χρειαζόμαστε τις απαραίτητες φυσικές καταβόθρες διοξιδίου του άνθρακα ε, που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο να επιτύχουμε την ε, ε, ουδετερότητα άνθρακα. Ε, στη θέρμανση, εκεί μπορούμε να χρησιμοποιούμε βιοκαύσιμα και να χρησιμοποιούμε ξύλο και να αντικαταστήσουμε με το ξύλο τις, τα καύσιμα που χρησιμοποιούν τώρα και είναι ένταση άνθρακα. μπορούμε να αντικαταστήσουμε πάρα πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούν στην κάψη και βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα. τώρα, στη γεωργία υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για να περιορίσουμε τις εκπομπές του θερμοκηπίου αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, στο πώς και το έδαφος μπορεί να δεσμεύσει τον άνθρακα. Σε αυτό το θέμα πρέπει να προχωρήσουμε, να επιτύχουμε βελτιώσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι οι διοκτήτες δασών και οι γεωργοί ε, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για όλα αυτά τα θέματα και γι' αυτό χρειάζονται υποστήριξη και ενθάρρυνση στη δουλειά τους. Και θέλω να υπογραμμίσω κυρίως τη σημασία της επιστήμης και της έρευνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να διαθέσει επιπρόσθετα κονδύλια στο μέλλον για την έρευνα και αυτά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα κύριε Επίτροπε έχετε το λόγο και έχετε και τον απαραίτητο χρόνο για να απαντήσετε σε όλα αυτά που ετέθησαν. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής που έθεσαν τις ερωτήσεις ε, πολύ ενδιαφέρουσες για αυτά τα θέματα ε, και που ενδιαφέρονται αλλά και κυρίως για την δράση τους στη διάδοση του μηνύματος και στην επαφή με τον κόσμο. Και βεβαίως ευχαριστώ για τα επενετικά σας λόγια. Είναι ε, πολλά υποσχόμενα αυτό για το μέλλον. Ξέρετε ότι οποτεδήποτε με καλέσετε ευχαρίστως επανέρχομαι. Ε, για να συζητήσω πάντοτε με ενθουσιασμό μαζί σας. Ε, ε, σήμερα συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει και σε τι θα πρέπει να εστιάσουμε. Εγώ θέλω να τονίσω κάποια πράγματα με το, για τα οποία θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ακόμα στην Επιτροπή ε, σε αυτό το πλαίσιο αλλά και με βάση τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπράφτση για το ενσαφή του δήλωση ότι η βιομηχανία είναι ε, έτοιμοι, είναι πλήρως ε, προσιλωμένη για αυτή την περίπλοκη προσπάθεια που χρειάζεται όμως πραγματικά για να μπορέσουμε να περάσουμε σε αυτή τη μετάβαση, ε, να επιτύχουμε μάλλον αυτή τη μετάβαση. Χρειάζεται βοήθειά μας στη βιομηχανία για την έρευνα και την καινοτομία. Ελπίζω πως αυτά τα νέα κονδύλια τα οποία θα δημιουργηθούν, το Ταμείο για τον Εξυγχρονισμό και το Ταμείο για την καινοτομία με βάση τα εισοδήματα από το πρόγραμμα ανταλλαγής εκπομπών, εμπορίας μάλλον εκπομπών, ε, θα βοηθήσουν σε αυτό. Αυτά εγκρίθηκαν ε, και προτάθηκαν μάλλον από την Κομισιόν και μάλιστα αυξήθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο και θα είναι ε, η μεγαλύτερη, τα μεγαλύτερα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να πάνε στην έρευνα βεβαίως και να περιλαμβάνεται εκεί οτιδήποτε έχει να κάνει με τους τομείς που χρησιμοποιούν πολύ ενέργεια και με οτιδήποτε έχει να κάνει με την απαλλαγή από τον άνθρακα. Θέλω να πω δύο λόγια γιατί έχουμε και ακούμε διάφορα νέα για προκλήσεις ε, όσον αφορά τον τομέα του Χάλιβα. Ε, μεγάλα προβλήματα και είναι πολύ, ευγεν... πολύ ε, δύσκολο θέμα και οι εργαζόμενοι στο Χαλιβουργία είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι και πάντοτε ανησυχούν όταν βλέπουν τόσο μεγάλες διακοιμάνσεις και επιτητικότητα στην αγορά. Συναντήθηκα και συζήτησα με τη συνάδελφο Σεσίλια Μάλστρομ που είναι υπεύθυνη και πρέπει να σας πω ότι πάνω από 20 άνθρωποι εργάζονται και ανάλογον την ε, σημερινή κατάσταση μελετούν τις εισρωές του Χάλιβα που φαίνεται πως δεν έρχεται μόνο από την Ασία αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου και αυτό αποδεικνύει ότι αν ε, υπάρχει πληθυντικότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, αν είναι σε απρόβλεπτος όπως ε, είναι ο μεγάλος μας ε, υπερατλαντικός εταίρος, αυτό έχει συνέπειες σε συγκεκριμένα στους ανθρώπους, σε πολίτες και μετά έχουμε ζητήματα τα οποία πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε και σας διαβεβαιώ ότι όντως ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία. Ο κύριος Ρούπκια αναφέρθηκε στη σημασία του ε, κοινωνικού διαλόγου. Να πω ότι και εγώ εκτιμώ πολύ το πώς γίνεται αυτός ο διάλογος στην Αυστρία, λειτουργεί και φέρνει και αποτελέσματα και αυτό πιστεύω ότι η ε, υψηλή ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου ε, είναι κάτι το οποίο είναι υποδειγματικό στην Αυστρία και έχει λειτουργήσει και ως παράδειγμα για άλλες χώρες. Προσπαθούμε να, ε, μιμηθούμε, να σας μιμηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί ε, χρειαζόμαστε αυτή, αυτό το διάλογο. Πρέπει λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι κάθε φορά να κάθονται στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων και να ζητούν από κοινού τι καλύτερε λύσει. Μόνο όταν αυτό ε, ε, συμβαίνει, έχουμε καλά αποτελέσματα και ακόμα και αν ε, δεν συμφωνούμε πάντοτε μεταξύ μας έχει τουλάχιστον γίνει σωστή προσπάθεια και, δεν, ε, και αποφεύγουμε δραματικές καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ περισσότερα προβλήματα. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως μαζί σας ότι όταν ο κόσμος βλέπει πώς ε, αποδίδουμε και όταν λέω αποδίδουμε σημαίνει ότι εμείς, εμείς δουλεύουμε ε, για εκείνους πολύ συχνά ε, στρέφονται προς εμάς και ξεπερνούν τους λαϊκιστές. Ξέρουν ότι αυτά που προτείνουν ε, δεν λειτουργούν, όμως ε, είναι πολλές φορές ελκυστικές οι προτάσεις αυτών των ανθρώπων και να εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε εδώ για τους πολίτες και ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε αποτελέσματα. Επίσης ε, και αυτά τα σχόλια που έκανε ο κ. Σπίντος για την εταιρική ευθύνη και είμαι ευτυχής που αυτά λαμβάνονται όλα ένα και περισσότερο υπόψη βλέπουμε τι είδους ενέργεια μπορεί αυτό να ε, παράγει, πόσο συμβάλλει στον κοινωνικό ιστό ή και στο περιβάλλον εκεί όπου ανοίγει νέα εταιρεία. Ο κύριος Χέμελινγκ ε, μας θύμισε ότι ε, εγκρίθηκε η πρόταση για την ενέργεια ε, Πρέπει όμως να παρακολουθούμε πιστά και να, βλέπω να φτάσουμε στο στόχο στο 25, το 30 ε, και έχουμε κάποια κράτη-μέλη που ε, ε, υστερούν όσον αφορά την ε, επάρκεια ενέργεια και τα λοιπά, ε, δεν είναι κακή ε, θέληση ή έλλειψη αποφασιστικότητας. Πολλές φορές σημαίνει έλλειψη χρηματοδότησης ή ανάγκη για πυρογνωμοσύνη, για βοήθεια, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη, η Ευρώπη των 28 θα προχωρά με τον ίδιο ρυθμό για να μπορούν οι πολίτες να δούνε τα πλεονεκτήματα. Κύριε Μάκινα, θα τα, σας τα πω εσάς σλοβακικά. Ε, για, μας, ε, εσείς μας τονίσατε ε, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ε, ε, αποκλήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και πρέπει να σας πω ότι όλο και συχνότερα όταν ταξιδεύαστε κυρίως στα νέα κρατημέλη ε, θα θυμάστε, θυμάται ο κόσμος καλά το τι συνέβη και το πώς, ε, ε, ε πώς ήταν, σε τι κατάσταση ήταν οι οικονομίες μας για να μην το πω 50% κάτω από το μέσο όρο του ΑΕΠ. Τώρα βρισκόμαστε κατά 80% έχουμε φτάσει στο μέσο όρο. Όμως όχι για το προσωπικό εισόδημα. Ενώ το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 30% το εισόδημα, τα εισοδήματα χοντρικά αυξήθηκαν μόνο κατά 10%. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να εξασφαλίσουμε την ισότητα για όλους. Ακόμα και όταν πρόκειται, ε, μάλλον κυρίως και όταν πρόκειται για τα εισοδήματα. Κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει να εξαλείψουμε και τις εντάσεις που βλέπουμε ε, στα κράτη-μέλη είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα των τιμών της ενέργειας, όπως μας θύμισε η συνάδελφος. Και τώρα ε, γι' αυτό κάνουμε και βαθύτερη ανάλυση του κόστους της ενέργειας. Ποια είναι η τιμή της παραγωγής, ποιο είναι το κόστος της παραγωγής και ποια είναι, ποιες είναι οι επιπλέον ε, ε, προσθήκες. Μπορεί να φτάσει δηλαδή σε κάποια κράτη-μέλη η τιμή και 60% από την τιμή της παραγωγής. Και αυτό είναι ερώτημα για όλους μας. Είναι δίκαιο να φορτώνεις με τόσους φόρους ένα βασικό ε, και απαραίτητο αγαθό. Να δούμε δηλαδή άλλα μοντέλα για το φορολόγηση της ενέργειας. Να συγκρίνουμε το κόστος της παραγωγής ενέργειας, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν φυσικά πολύ πιο δίκαιο και θα ελάφρυνε τους πολίτες. Ε, η κυρία Ντομπρόφσκα μας θύμισε ότι αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα ε, για το μέλλον ή να τα προλάβουμε, θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Και πιστεύω πως το ερώτημα της ήταν σαφές και περιλάμβανε σημαντικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι πώς θα συμπεριλάβουμε στις εμπορικές μας συμφωνίες μια αναφορά για να καλύψουμε την ένταση. Την ένταση όχι μόνο από τη γεωργία, από την ε, αυτοκινητοβιομηχανία, από τη χαλιβουργία, για, ας πούμε, για ένα τόνο που παράγεται στην Ευρώπη χρειάζεται 1,8 τόνος ε, του άνθρακα. Ενώ αν δούμε το χάλιβα εκτός Ευρώπης συχνά φτάνει στο 3 ή στο 4 τόνους ε, άνθρακα ε, για το ίδιο προϊόν. Οπότε θα πρέπει να ζητήσουμε από τις αρχές μας να μην Μάλλον, ναι, μεν οι δημόσιε αρχέ επιλέγουν πάντοτε την καλύτερη τιμή, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο. Πρέπει να φροντίζουμε ώστε όλε οι επενδύσει που κάνουμε για την καθαρότερη και πρασινότερη παραγωγή στην Ευρώπη θα αποδώσουν και ότι οι παραγωγοί μας δεν θα τιμωρηθούν επειδή παράγουν με καθαρότερο τρόπο και να βγαίνουν από την αγορά ε, ε, λόγω ε, προϊόντων που έρχονται από άλλες αγορές όπου αυτοί οι κανόνες δεν τηρούνται. Ο κύριος Φουρνιέ τώρα τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε στο μυαλό μας την δικαιοσύνη, την ισότητα στην ενεργειακή μας πολιτική και πώς αυτό επηρεάζει τις διάφορες περιφέρειες. Ε, η... Τα νέα που μας στάνουν είναι ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πως κοινωνικά, πολιτικά αλλά και ανθρωπίνως είναι σημαντικό να δείξουμε πώς ε, μας ενδιαφέρει, πώς θέλουμε να βοηθήσουμε και πώς ξέρουμε και τι θα κάνουμε. Γι' αυτό και η ατμόσφαιρα που επικρατεί για αυτό του είδους συνεργασία είναι καλή και επιβεβαιώνω ότι χάρη στο Ευρωκοινοβούλιο και συγκεκριμένα χάρη στο Γέρζι Μπούζεκ έχουμε τώρα μία πρόταση για μία ειδική γραμμή του προπολογισμού 5 εκατομμύρια ε, νομίζω ευρώ είναι ε, για να ε, φιερωθούν στις περιφέρειες όπου ακόμα χρησιμοποιείται πολύ εντατικά ο άνθρακας να δουν αυτές τις περιφέρειες πως υπάρχουν οράματα και τα project τους μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Η κυρία Ματζόλα λέει πολύ σωστά ότι οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας δύσκολα μπορούν να μπουν με νέο τρόπο σε όλα τα νοικοκυριά. Μπορούμε όμως να ενισχύσουμε τα ηλεκτρικά οχήματα για παράδειγμα εφόσον τα δίκτυά μας γίνουν περισσότερο ευφύ. Οπότε και αυτό είναι ένα σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος. Έχουμε πρώτα απ' όλα εγκρίνει και χρηματοδοτικά τα πρώτα εφή δίκτυα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε να έχουμε περισσότερη κάλυψη και οικονομικά ώστε τα δίκτυά μας να γίνουν γρήγορα περισσότερα εφή. Και δύο σχόλια ακόμα από την κυρία Μαέροβα και του Σίμον Κιάνεν που αναφέρθηκαν στην ανάγκη επικοινωνίας. Συμφωνώ με τη συναδερφό μου, τη συμπατριώτησά μου, ότι ο δημόσιος διάλογος με συμμετοχή του κοινού είναι ζωτική σημασίας. Είναι αναπόφευκτο και πιστεύω ότι δεν κάνουμε αρκετά για να καταλάβει ο κόσμος τι προσπαθούμε να πετύχουμε, γιατί έχουμε καταλήξει στις προτάσεις που έχουμε καταλήξει για παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι πιο έντονη η επαφή αυτή, να είμαστε περισσότερο ορατοί, να προβληθούμε στα κοινωνικά δίκτυα και να φροντίσουμε να συμμετέχουν και οι νέοι να ενημερώνονται και οι νέοι για το τι κάνουμε, να μας καταλάβουν. Έτσι θα υποστηρίξει ο κόσμος περισσότερο τις προσπάθειές μας. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντικό για την νεολαία. Τώρα θα ακούσετε, φαντάζομαι, με ικανοποίηση ότι οι φυσικές καταβόθρες, ε, άνθρακα και όλα τα άλλα που συζητάμε αποτελούν αντικείμενο του νέου αυτού ταμείου για την ε, ε, βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή ανανέωση. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε όλα αυτά τα σχέδια τα οποία έχουν προτείνει οι Φιλανδοί. Τώρα, επειδή είμαι από την ε, Σλοβακία, θα σας πω κάτι που έχει σχέση και με την Φιλανδία. Ήμασταν πρωταθλητές στο χόκι. Η Φιλανδία πάντα τα καταφέρνει, έχει πάρα πολλούς υποστηριχτές, γιατί όπως ξέρετε το φιλανδικό όνομα αρχίζει από S. Φώναζε λοιπόν το γήπεδο Σουόμι, Σουόμι. Όμως χαιρόμαστε που θα μπορέσετε να συνεχίσετε να είσαστε πρωταθλητές. Ευχαριστούμε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς κύριε Σεύκοβιτς, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για το ότι ήρθατε εδώ και για το ότι ξεκινήσετε το διάλογο με μας. Νομίζω ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στον τομέα της ενέργειας δείχνει με απόλυτη σαφήνεια το τι υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η Επιτροπή έλαβε μία σαφή εντολή πριν από πέντε χρόνια και εσείς είσαστε ο πρωτοπόρος, ε, εσείς είσαστε εκείνος που αγωνιστήκατε κάθε μέρα πάντα με φοβερές διπλωματικές ικανότητες, χαμογελώντας, αναζητήστε λύσεις και διαπραγματευτήκατε με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους, με όλους τους ε, θεσμούς ε, και με τα 28 κρατημέλη για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο έτσι ώστε να θεσπίσετε νομοθετικές ε, ρυθμίσεις. Αυτή είναι η κληρονομιά που αφήνεται πίσω σας και τα επόμενα χρόνια κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη σημασία αυτής της ε, κληρονομιάς. Η αφαίρεση του άνθρακα από την Ευρώπη, αυτό είναι το, η βασική πρόκληση για τα επόμενα έτη. Θα επηρεάσει αναμφισβήτητα τον κόσμο των επιχειρήσεων, μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις ε, και βέβαια και μεγάλη ευκαιρία και κίνδυνος για τις επιχειρήσεις. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ε, εργαζόμενους, μεγάλη ευκαιρία, όπως είπα, αλλά και μεγάλος κίνδυνος. Και επίσης ε, θα είναι και μεγάλος κίνδυνος για αυτά που συζητάμε εδώ, που είναι ότι δεν θέλουμε να χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Ε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς που μας ανταγωνίζονται Το είδαμε στου υπολογιστέ. Εγώ έρχομαι από την Ιταλία. Ο Ολιβέτη είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Δεν πρέπει να χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μα. Ε, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να χάσουμε την υποστήριξη και τη συμμετοχή των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να χάσουμε έδαφος και την ε, εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Το θέμα είναι ε, το πώς θα μπορέσουμε με βιώσιμο τρόπο να περάσουμε το κόστος αυτής της ε, μετάβασης, πώς θα το μετακυλήσουμε στις τιμές. Αυτό είναι η βασική πρόκληση των επόμενων ετών. Το σημαντικότερο είναι να είμαστε ε, πολύ συγκεκριμένοι. Σας ευχαριστούμε και πάλι και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ξανά επανεκφράσω την επιθυμία μας να ε, ξαναέρθετε εδώ ή κάπου αλλού ως μέλος της Επιτροπής με ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα προκύψει μετά από όλες τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Θα ολοκληρώσουμε σε λίγο την Ολομέλεια, αλλά προηγουμένως πρέπει να ψηφίσουμε και να δούμε και τις τροπολογίες της ε, έκθεσης αυτής, στρατηγική για την μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πέντε τροπολογίες που έχει εγκρίνει και ο εισηγητής και ο συνεισηγητής από ό,τι έχω καταλάβει. Σωστά. Συμφωνείτε όλοι. Τότε ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Μπορείτε να ψηφίσετε. Le vote est 151 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Εγκρίθηκε λοιπόν η έκθεση αυτή συγχαρητήρια στον εισηγητή και τον συνεισηγητή. Και τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, πρέπει να εγκρίνουμε την ημερομηνία της επόμενης ε, Συνόδου Ολομέλειας, που θα είναι 17 και 18 Ιουλίου στο κτίριο Σαρλεμάνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι ομάδες μπορούν να συνδυάσουν στις 17 του μήνα από τις 9 το πρωί. Την ίδια μέρα στις 2.30 θα αρχίσει η Ολομέλεια και θα συνεχίσουμε τις εργασίες της Ολομέλειας την επόμενη μέρα στις 18 από τις 9. Ε, καλείται το σώμα να εγκρίνει τις ημερομηνίες αυτές. Συμφωνείτε? Ωραία. Καλή επιστροφή στις χώρες σας και θα τα πούμε στην επόμενη Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος.